και τα σχετικά κείμενα είναι στη διάθεσή σας, υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, τα πρακτικά εγκρίνονται. Αξιότιμοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της συνάντησης κορυφής της ζώνης του ευρώ στις 11 Μαρτίου. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ζούμε μια περίοδο όπου η ιστορία επιταχύνεται. Ένας άνεμος ελευθερίας πνέει και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που σπέβδω να σας ανακοινώσω ότι η Επιτροπή ενέκρινε την βοήθεια για τις χώρες της Μεσογείου στην διάρκεια της μετάβασης για να δοθεί νέα όθηση στην μεσογειακή μας σχέση, στις σχέσεις γειτονίας. Αυτό θα εγκριθεί και την επόμενη Παρασκευή. Οι νέοι στις χώρες της Βορειού Αφρικής διαδηλώνουν κατά της απολυταρχίας Είμαστε μάρτυρες ενός αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία. Αν και η κατάσταση είναι πολύπλοκη και παρουσιάζει γενείς προκλήσεις, εμείς ε, δεν πρόκειται να μισούμε τα λόγια μας. Είμαστε με αυτούς που διεκδικούν την πολιτική τους ελευθερία και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν θα αμφιταλαντευτούμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα καθεστώς το οποίο Βάλει κατά του λαού του δεν έχει θέση στον κόσμο αυτόν. Προτείνουμε στους λαούς της Βορείου Αφρικής μια σχέση εταιρική, μια σχέση συνεργασίας βασισμένη στους δημοκρατικούς θεσμούς, συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και την αλληλέγγυη ανάπτυξη. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Το να πούμε όμως όχι, να προστρέψουμε το βλέμμα δεν συνάδει με την δημοκρατία. Ο δρόμος προς τη δημοκρατία δεν είναι ποτέ εύκολος. Πολλές φορές είναι δύσκολο, απαιτητικό, όμω η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο πλευρό αυτών που επιδιώκουν την πολιτική του ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κυρίε και κύριοι, την Παρασκευή 11 Μαρτίου συνεδριάζει του Ευρώ στο ανώτερο επίπεδο. Η κρίση μας έδειξε σε ποιο βαθμό είναι αλληλένετες οι οικονομίες μας. Η κρίση κατέδειξε και μερικές διαρθρωτικές αδυναμίες. Γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε να ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση. Η Κομισιόν από καιρού υπεραμείνεται της ανάγκης περαιτέρω συντονισμού των εθνικών οικονομιών και της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Προτείνουμε πυλώνας της ΟΝΕ να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Και το είχαμε υπογραμμίσει αυτό στην έκθεσή μας για τα δέκα χρόνια του ευρώ. Η είναι όμως ότι κάποιοι ηγέτες δίστασαν. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση αποτελεί αδύρυτη αναγκαιότητα. Μας το επιθυμίζουν και αγορές. Υπό την Προεδρία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταλήξαμε σχεδόν ομόφωνα υπέρ μια ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Οι προτάσει είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για το Συμβούλιο. Κατά τα άλλα συμφωνήσαμε για την υλοποίηση ενό Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει τι σχετικέ αποφάσεις και που θα συμπεριλάβει όχι μόνο τι δημοσιονομικέ πολιτικέ, αλλά και τι οικονομικέ πολιτικέ και τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό της οικονομικής, δηλαδή της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης, προέκυψε πρόσφατα η ιδέα ενός συμφώνου ανταγωνιστικότητας, για να κάνει δηλαδή η Ευρώπη επιπλέον προσπάθειες στο πλαίσιο των εθνικών αρμοδιοτήτων για να γίνουμε ως Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Είναι αλήθεια ότι εάν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς είμαστε αλληλοεξαρτητοί, αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την ζώνη του ευρώ. Τώρα, οι διαφορέ στην ανταγωνιστικότητα είναι πρόβλημα για χώρε οι οποίε μοιράζονται το ίδιο νόμισμα. Η ανταγωνιστικότητα και η σύγκληση είναι λοιπόν ουσιώδει παράγοντε για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα τη ζώνη του ευρώ και τούτο για το καλό τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι η ιδέα αυτή γέννησε ανησυχίε, φόβου για μια ζώνη, για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ορισμένοι φοβήθηκαν ότι μπορεί να ακυρώσουμε την ανάκαμψη. Άλλοι ότι αμφισβητείται η κοινωτική προσέγγιση. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι θεμητά και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις χωρίς αφιταλαντεύσεις. Πρόκειται για ζητήματα αμοιβέ εμπιστοσύνη. Κυρίε και κύριοι, και εγώ εξεπλάγιν που χρειάστηκε να υπενθυμίσω στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο στις 4 Φεβρουαρίου ότι κάθε πρωτοβουλία στον τομέα αυτών πρέπει φυσικά να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνθήκης. Στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, παραθέτω, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα λάβουν συμπληρωματικά μέτρα με στόχο να προσδώσουμε νέα ποιότητα στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει ακόμη περισσότερη σύγκληση χωρίς να φυγεί η εσωτερική αγορά. Χάρηκα πολύ επίσης που προσθέσαμε στα συμπεράσματα ότι αυτές οι πρόοδοι, τα βήματα πρέπει να γίνουν συμφώνως προς την συνθήκη. Ε, εννοείται βεβαίω, αλλά καλό είναι μερικέ φορέ να το λέμε, ακόμα και αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Δόθηκε λοιπόν εντολή στον πρόεδρο του Συμβουλίου, σε συνεργασία με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη να προχωρήσει για να εξεύρει τα μέσα με τα οποία θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Αυτέ οι διαβουλεύσει έδειξαν σαφώ ότι εν γέννη τα κράτη-μέλη είναι υπέρ τη κοινοτική προσέγγιση. τα μέλη, θα ήθελα να είμαι σαφή όσον αφορά τι ε, αρχέ, οι οποίε κατά τη γνώμη τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, πρέπει να τηρηθούν στο πλαίσιο αυτού του συμφώνου ανταγωνιστικότητα. το οποίο θα ήταν καλύτερο να το αποκαλούμε σύμφωνο σύγκληση και ανταγωνιστικότητα, γιατί ακριβώ σκοπό μα είναι να μειώσουμε τι αποκλήσει μέσα στη ζώνη του ευρώ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Η πρώτη αρχή είναι ότι το σύμφωνο αυτό πρέπει να συνάδει με την συνθήκη στο πλαίσιο του υφισταμένου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης. Μόνο έτσι θα είμαστε βέβαια για, την κοινοτική, για, τον κοινοτικό χαρακτήρα της προσέγγισης. Η εμπειρία μας με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δείχνει ότι μόνο με την κοινοτική μέθοδο, με την κοινοτική προσέγγιση μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αποδεκτά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο θα είναι δεσμευτικά. Το σύμφωνο επίση πρέπει να κάνει σεβαστό τον ρόλο τη Κομισιόν για λόγου αντικειμενικότητα, για λόγου εσωτερική αγορά, για λόγου σεβασμού του κοινωτικού κεκτημένου και για λόγου συνοχή μεταξύ των μέτρων εντό τη Ευρωζώνη και αυτών που λαμβάνονται γενικότερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα τονίσω επίση τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτήρηση, επίβλεψη αυτού του μηχανισμού. Θα τηρούμε ενήμερο βεβαίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σύμφωνο επίση πρέπει να είναι ανοιχτό και σε άλλα κράτη-μέλη, τα οποία ενδεχομένω θέλουν να συμμετάσχουν, τα οποία δηλαδή δεν είναι μέλη τη ζώνη του ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην δημιουργήσουμε ξεχωριστέ κατηγορίε μελών εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν θα ήταν συμβατό με τις αρχές μας. Για να δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, ένα τέτοιο σύμφωνο που απαιτεί εθνικά μέτρα, πρέπει να υπάρχει προσθεμένη αξία φυσικά στα όσα έχουμε ήδη κάνει με τις προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Να σας υπενθυμίσω ότι βάσει του άρθρου 121 της συνθήκης τα κράτη-μέλη οφείλουν να συντονίζουν τις εθνικές τους οικονομικές πολιτικές. Γι' αυτό προσεγόντας να μην στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά. Ίσα ίσα να την βελτιώνουν. Επιπλέον πρέπει ο κοινωνικό διάλογος να προάγεται ταυτόχρονα και να επιδιώκονται στόχοι όπως η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας όπως λέει και η Agenda 2020. Η ανταγωνιστικότητα είναι απολύτω απαραίτητη για τι χώρε μα. Είναι προαπαιτούμενο για την δημιουργία αναπτύξη και θέσεων εργασία. Γι' αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλίζουμε ότι αυτό το σύμφωνο θα παρέχει πραγματικά προστιθέμενη αξία και δεν θα μα απομακρύνει από του βασικού μα στόχου, τη ανάπτυξη δηλαδή και των νέων θέσεων εργασία. Γι' αυτό τονίζω συνεχώ την αξία τη ανάπτυξη και μάλιστα τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι στην καρδιά τη Ατζέντα 2020. Και να τονίσω και την κοινωνική πτυχή. Οι προσπάθειε πρέπει να κατανέμονται ισομερό. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή μελετά προτάσεις όσον αφορά την φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εάν απαιτείται δημοσιονομική εξυγίανση για την πρόοδο, απαιτείται και επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Να μην ξεχνούμε επίση ότι το σύμφωνο είναι μέρο μόνο τη συνολική μα απάντηση για να εξασφαλίσουμε να προστατεύσουμε την σταθερότητα τη ζώνη του ευρώ. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα και άλλε απαντήσει για να διορθώσουμε της ελλείψης του μηχανισμού, του σημερινού μηχανισμού σταθερότητας. Πρέπει να πορευτούμε προς έναν μόνιμο μηχανισμό το 2013 και να τον εφαρμόσουμε τους επόμενους μήνες θέλοντας και πιο αυστηρούς κανόνες για τις τράπεζες, για περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Το σύμφωνο θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο εάν ερμηνευθεί ως μέτρο στο πλαίσιο, όπως είπα, και άλλων πρωτοβουλειών και μέτρων για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Θα μπορούσε να συμβάλλει σε περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, εάν είναι συνεκτικό και συμβατό με το κοινοτικό σύστημα διακυβέρνησης. Γι' αυτό απαιτείται λοιπόν η κοινοτική προσέγγιση. Έτσι, θα έχουμε να συνεισφέρουμε με προσθεμένη αξία μάλλον έναν πυλώνα στην οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θέλει η Κομισιόν, αυτό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αφιστούμε ε, κόπον για την επιτυχία αυτού του νέου συμφώνου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και περνούμε τώρα στους ομιλητές εξ των ομάδων. Ο πρώτος ομιλητής εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ντόλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι δίδαγμα λαμβάνουμε από την χρηματοοικονομική κρίση. Από τον Παγκόσμιο Πόλεμο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι λαοί έπρεπε να συνεργάζονται και όχι να ασφάζονται. Από την πτώση του τείχου του Βερολίνου μάθαμε ότι μπορούσαμε να επανενώσουμε την ήπειρό μα γύρω από αξίε δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική οικονομία τη αγορά. Από την τρομοκρατική επίθεση τη 11η Σεπτεμβρίου μάθαμε ότι πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Από την σημερινή κρίση, τι θα έπρεπε να διδαχθούμε. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να πάψουν να θεωρούν ως ταμπού την, ε, συνεργασία στους φορολογικούς, δημοσιονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Ένα τμήμα του δρόμου το ακολουθήσαμε. Φέτο ξεκινήσαμε τον συντονισμό των 27. Ήδη ο συντονισμός αυτός σε δημοσιονομικό επίπεδο είναι ένα, μια επανάσταση. Μάθαμε να υιοθετούμε κανόνες για να κάνουμε πιο ηθική την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η ομάδα μου ζητά να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου πριν το καλοκαίρι για μια ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Η ομάδα μου ζητά επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειες συντονισμού για την κοινωνική και οικονομική και φορολογική διάσταση στο πλαίσιο του συμφώνου μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα ωστόσο και να εξασφαλίσουμε ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και οι Επιτροπή θα ασκούν όλα τα δικαιώματα που τους ανήκουν στον τομέα αυτό. Στηριζόμαστε σε αυτό στον πρόεδρο της Επιτροπής. Η ομάδα του ΕΛΚ καλωσορίζει και υποστηρίζει τις προτάσεις αυτές, όπως το έκαναν και στο Ελσίνκι οι εθνικοί ηγέτες του κόμματος. Κυρίες και κύριοι, πώς να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι παρότι υπάρχει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στα μέσα Ιουλίου κάθε χρόνο, τα περισσότερα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεχίσουν να, δια... να δαπανούν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Η υπερχρέωση των κρατών πώ θα μπορούσε να είναι πιο αποδεκτή από την ε, υπερχρέωση των επιχειρήσεων ή των νοικοκυριών. Η κρίση δημιούργησε κατάργηση θέσεων εργασίας, οικογενειακά δράματα. Από αυτό πρέπει να διδαχθούμε και να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Πρώτο μάθημα. Να μην αντιμετωπίζουμε ελαφρά την καρδία τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη ανεξάρτητα από το μέγεθός τους για την τήρηση των δημοσιονομικών ορίων. Δεύτερο μάθημα. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο εάν οι κανόνες σε δημοσιονομικό, σε φορολογικό και ε, κοινωνικό επίπεδο είναι συγκρίσιμοι, τουλάχιστον συγκρίσιμοι, κάτι που δεν συμβαίνει. Τρίτο μάθημα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα μηχανισμό σταθερότητα για την προστασία τη κοινωνική οικονομία τη αγορά μα. Τέταρτο και τελευταίο μάθημα. Μέσα στη θύελα η Ευρώπη στέκει. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ενισχύεται. Οι, οι Αμερικανοί και οι Ιαπωνέζοι εταίροι μα έχουν πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση χωρί να ανισχούν ιδιαίτερα. Πρέπει να το πούμε αυτό. σω αυτό να μην ισχύσει για πάντα. Από πλευρά μα είναι η στιγμή να εξηγιάνουμε την οικονομία και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, να δουλέψουμε για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Ντόλ. Εξ ονόματος της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Μάρτιν Σούλτσε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι λίγοι βουλευτές, εδώ και εβδομάδες συζητούμε για ένα έγγραφο των ε, Σαρκοζή και Μέρκελ που δεν υπήρχε επί του μη υφισταμένου κειμένου όμως ε, δόθη συνέντευξη τύπου και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και είχε και περιεχόμενο συγκεκριμένο το οποίο ε, δεν γνωρίζομαι ε, και δεν, το περιεχόμενο δεν θα γίνει ε, πραγματικότητα. όλα αυτά όμως υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένα συμπεράσματα σε σχέση με το μηχανισμό διάσωσης. Δηλαδή αυτή ήταν η εξέλιξη. Η κατάσταση είναι καυκική. Η διάσωση του ευρώ δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ε, μου άρεσε ο λόγος σας κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής διότι οι κοινωνικές ανισορροπίες παρουσιάστηκαν σωστά. Εξεπλάγει λίγο γιατί η Ομοσπονδιακή Γερμανία με την καγκελάριό της ζητεί όπως και ο κύριος Σαρκοζή μέτρα τα οποία δεν έχει λάβει η Γερμανία με αυτή τη μορφή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός, όλοι οι προϋπολογισμοί ε, θα πρέπει να περικοπούν. Τι έχει γίνει ε, κατά το παρελθόν. Ε, έχουν εφευρεθεί πριν τα οποία ανάλογα σταθεροποιούν τους πάσχοντες τομείς. Βλέπε αυτοκίνητο βιομηχανία. Έτσι αντιμετωπίστηκε βέβαια ε, εντελώς παρεμβατικά ε, το πρόβλημα στη Γερμανία. Γιατί με τις ιδιαιτερότητες τους το καθένα να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν το ίδιο. Το, η ε, κατεβάζει την Ελλάδα κάτω από τη Λευκορωσία και την Αίγυπτο. Αυτό έγινε πρόσφατα. Και αναρωτιέται κανείς ε, είναι δυνατόν ή έχουμε τρελαθεί ακόμη και κάτω από το Βιετνάμ και τρεις μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής γίνονται αυτά. Τρεις μέρες πριν από μια Σύνοδο Κορυφής ε, γίνονται τέτοια πράγματα. Η Μούντις τι λέει, αξιολογούμε προς τα κάτω διότι η χώρα ε, δεν μπορεί πλέον να κάνει επενδύσεις και δεν μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη. Ε, συζητάμε λοιπόν για το haircut. Το haircut, το κούρεμα, πιστέψτε με, το ξέρω δεν λύνει τα προβλήματα. Και στο τέλος ε, τι θα γίνει. Η πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας θα πρέπει να αυξηθεί λέγοντας ε, ότι θα ε, ε, σταματήσουν οι παραγραφές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει απαραίτητος να παρέμβει ένας μηχανισμός διάσωσης. Ένα τέτοιο σύμφωνο ε, θεωρητικά είναι σωστό, αλλά στην πράξη χωλαίνει, διότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολύ συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες για την αποκατάσταση μιας ισορροπίας. Με βάση αυτά που είπατε, ε, νομίζω ότι το σύμφωνο πηγαίνει προς τη σωστή πορεία. Γι' αυτό λέω ότι η πρότασή σας είναι σωστή. Δεν θα μιλήσω πολύ για το θεσμικό ζήτημα. Σε θεσμικό επίπεδο η προσέγγιση δεν ήταν σωστή. Θα πρέπει να δούμε ε, τις βάσεις ε, των ε, επιχειρησιακών μας προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να υπάρχει έδραση στους θεσμούς, ούτως ώστε να υφίσταται και δημοκρατική νομιμοποίηση. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε άσχημα, ε, ακολουθήσαμε σε ολισθηρό δρόμο, τώρα προχωράμε σωστά, γίνονται ορισμένες ε, σωστές προτάσεις που φαντάζομαι ότι θα ε, συμφωνήσουν και στη Γερμανία. Ε, θα έχουμε δηλαδή μια, ένα σύμφωνο για το ευρώ. Ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αρκετά καλά. Ευχαριστούμε τον Μάρτιν Σούλτσε και τώρα η ομάδα των φιλελευθέρων δημοκρατών. Τρία λεπτά ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ. Καταρχάς νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ε, μετά από χρόνια κατά τα οποία δεν είχαμε δεχθεί την ιδέα της Οικονομικής Ένωσης, τελικά δεχόμαστε την έννοια της Οικονομικής Ένωσης δίπλα στην νομισματική. Δεν είναι και καμία πολύ εξελιγμένη ιδέα, μόνο ο ως Φάρατς και κάποιοι άλλοι δεν το θέλουν. Αλλά κύριε Πρόεδρε, ο όρος που χρησιμοποιείται είναι κακός. Σύμφωνο. Τι σημαίνει σύμφωνο. Σύμφωνο είναι συμφωνία μεταξύ κρατών. Δεν θέλουμε συμφωνία μεταξύ κρατών. Θέλουμε μια κοινοτική πράξη. Μια πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ένα σύμφωνο μεταξύ των κρατών μελών που εξορισμού είναι διακυβερνητικό. Άρα ο όρο δεν είναι σωστός. Δεύτερον, η μέθοδος. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι κάτι διακυβερνητικό. Ο διακυβερνητισμό ουδέποτε λειτουργήσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική τη Λισαβόνα ήταν διακυβερνητική. Απέτυχε. Το σύμφωνο σταθερότητα, όταν η Γαλλία και η Γερμανία δεν το τήρησαν το 2003 και 2004, δεν τήρησαν του κανόνε του συμφώνου, αποδείχθηκε εκ νέου ότι η διακυβερνητική μέθοδο δεν λειτουργεί, δεν είναι σωστή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινοτική μέθοδο. Και τρίτον, Νομίζω ότι αυτό που υπάρχει επιτάπητος κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής δεν είναι επαρκές. Χρησιμο, μάλλον προσανατολίζεται σε συγκεκριμένα μέτρα. Το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας των κυρίων, ε, της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή είναι πολύ ε, εξειδικευμένο. Το συνταξιοδοτικό, λένε, η ηλικία συνταξιοδότηση ε, να αυξηθεί. Μα δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν τα χρόνια, υπάρχουν οι εισφορές είναι αν υπάρχει όχι δεύτερος πυλώνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι έξι συγκεκριμένα μέτρα σε ένα διακυβερνητικό σύμφωνο που δεν θα λειτουργήσει ή δεν θα υπάρξει ποτέ, αλλά μία εκτεταμένη οικονομική διακυβέρνηση που θα καλύπτει συνταξιοδοτικά συστήματα, αγορά εργασία, μισολογική πολιτική, φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποφασίζεται από την Επιτροπή που θα αποφασίζεται από την Επιτροπή και μέσω της ενός κώδικα σύγκλησης παρέχεται στα κράτη μέλη ζητώντας τους να εφαρμόσουν τους κανόνες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κώδικα σύγκλησης και το συντομότερο δυνατό. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι απλό. Είδα το κείμενο της 25ης Φεβρουαρίου. Το δικό σας και του κ. Βαν Ρομπάι. Τώρα είναι καιρός να ξεκινήσει την πρωτοβουλία τη δική της Επιτροπή. Μπορείτε να το κάνετε τώρα. Έχετε χρόνο τις επόμενες εβδομάδες να προετοιμάσετε αυτό το κοινοτικό κείμενο για την η οικονομική σύγκληση και διακυβέρνηση και να καταθέσετε την πρότασή σας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εμείς θα αποφασίσουμε και θα σας υποστηρίξουμε. Προς το παρόν, ωστόσο, η Επιτροπή έχω την εντύπωση ότι παρακολουθεί το κείμενο της 25ης του και βλέπω, τι βλέπω, μόνη την παρακολούθηση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Δεσμεύσεις που λαμβάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Μα δεν θα λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι τα κράτη ή πρωθυπουργοί που θα ελέγχουν τους εαυτούς τους. Ουδέποτε λειτουργήσε, ούτε τώρα θα λειτουργήσει. Και τελευταία παρατήρηση, νομίζω ότι είναι καιρός, πρόεδρε της Επιτροπής, να υπάρξει μία πρωτοβουλία το συντομότερο δυνατόν για τους μηχανισμούς κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για, για τις τράπεζες μια και είστε υπεύθυνο, εσεί πρέπει να το κάνετε κύριε Πρόεδρε, γιατί είστε υπεύθυνο για την σχετική εποπτεία. Ευχαριστώ και μπορείτε να ξεκινήσετε. Εξ ονόματο της ομάδα των Πρασίνων για 3,5 λεπτά η Ρεμπέκα Χάρμ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι υποχρεωμένη να πω τίποτε πια για την επώδυνη ιστορία ε, αυτού του συμφώνου, διότι ακούσαμε ότι δεν υπάρχει το έγγραφο, αλλά στους διαδρόμους της Βρυξέλλες το Συμβούλιο διενέμετο παντού. Είχα πει ότι κάποια στιγμή ότι είχε όψιμα σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά, ε, κατά αναλογία προς τα όψιμα κομμουνιστικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με το πώς ε, αντιμετωπιζόταν η πραγματικότητα στα κτίρια του Συμβουλίου είναι κάτι παραπάνω από νομισματική κρίση αυτή. Εδώ και μήνες στην Ευρώπη βλέπουμε μια κρίση ικανοτήτων των εθνικών κυβερνήσεών μας να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη ενώπιον της κρίσης και να συμφωνήσουν από κοινού μέτρα εξόδου από την κρίση. Ε, αν ε, αποφασιστεί ο μηχανισμός, όπως και αν δημιουργήθηκε, θα έχει γίνει ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να πω όμως ότι αν κοιτάξουμε σήμερα την Ελλάδα βλέπουμε πόσο απατηλό ε, μπορεί να είναι το ότι πιστεύουμε ότι ξεπεράσαμε την κρίση ήδη. Διότι φαίνεται στη χώρα αυτή ότι τα μονόπλευρα μέτρα που προσανατολίζονται μόνο στην εξοικονόμηση και τη λιτότητα δεν έχουν αποτέλεσμα. Η χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύει. Όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα μειώνει τα έσοδα τόσο δραστικά θα πρέπει να ε, γνωρίζει ε, ποιες θα είναι άλλες πηγές εσόδων και θεωρώ ότι και εν ώψη αυτής της συνόδου και εν ώψη της αμέσως επομένης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε την ε, άρνηση που υπάρχει από τη Γερμανία για τη συμφωνία σε μέτρα και διευκολύνσεις. Θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, να καταλάβουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Η οικονομική πολιτική και η οικονομική ένωση απαιτεί μέτρα εξυγίανσης αλλά και την ε, αλληλεγγύη στην πράξη. Και εκεί η Ελλάδα ε, θα έχει περισσότερα να περιμένει από αυτά που έλαβε μέχρι τώρα. Μετά τον Μάρτιν Σούλτς και τους προλαλήσαντες ε, και εξ ονόματος των συναδέλφων που ασχολούνται με μήνες για το θέμα αυτό θα ήθελα να πω ότι η κοινοτική μέθοδος δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ε, σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς στις Βρυξέλλες. Αυτό χρειάζεται ούτως ώστε οι πολίτες από την Ελλάδα μέχρι τη Δανία, τη Γερμανία, και την Ισπανία να μας εμπιστεύονται. Εάν ε, θέλουμε να λειτουργήσουμε ως closed shop, ε, όπως αναφέρεται ε, και στα πλαίσια του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας, τότε θα χάσουμε την αξιοπιστία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι που διακυβεύεται όλο και περισσότερο σούσεις της κρίσεως. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε το Συμβούλιο αυτό να επιδείξει μεγαλύτερη λογική από ό,τι μέχρι τώρα. Τέλος, ε, ε, μιλήσατε για την αηφόρο βιώσιμη ανάπτυξη κύριε Μπαρόζου. Ε, γιατί ένας επίτροπος για την ενέργεια λέει σήμερα ότι η προστασία του κλίματος ε, σημαίνει ε, αποβιομηχάνηση. Ο Γερμανός Υπουργός Περιβάλλοντος ήταν στις Βρυξέλλες πριν από δύο εβδομάδες και παρουσίασε μία μελέτη που δείχνει 6 ε, εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας ε, αν θέσω μέσα στο 30% το στόχο του περιβάλλοντος. Ε, αύξηση λοιπόν της απασχόλησης μέσα από τα σωστά μέτρα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών της Ευρώπης για ένα λεπτό η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ. Σε μια στιγμή κρίσης πρέπει να υπάρξει ταχεία δράση. Είναι σαφές ότι η Ευρωζώνη δεν έχει βγει από την κρίση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να ανάλαβει κανεί έξυπνη δράση. Η Μεγάλη Βρετανία επανέφερε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με μείωση του εθνικού χρέου και αλλαγέ ε, και μείωση του ελλείμματο, κάτι που είχε συνέπειε. Οι διαδικασίε του Κοινοβουλίου δεν μα επιτρέπουν να λάβουμε γρήγορε αποφάσει. υπάρχουν προτάσει Ευρωβουλευτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια στην Ιρλανδία, κάποιοι από εμά ε, δανείσαμε, αυτοί που δανείσαμε άλλες χώρες αξίζουν επιτόκια που αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο και τα χρήματά του πίσω. Εγώ θα έπρεπε, προτείνουμε να υπάρχει ένα μπόνους όταν αποπληρώνεται νωρί το χρέο. Στο πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στο δικό του εθνικό προπολογισμό. Προτείνω το ίδιο να συμβεί και για, τους, ε, και για τη συνεισφορά των ε, φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή στο ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ελπίζω οι εθνικέ κυβερνήσει παρά την κρίση να ακούσουν τι προτάσει μα και να δουλέψουμε με συνολικά και αθληστικά με επικοδομητικό τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα από, για την Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά ο κύριος Μπίσκη δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο. Με χαρά σημείωσα ότι το κοινωνικό ζήτημα ε, το αναδείξατε και τάσεστε υπέρ των κοινωνικών ισορροπιών είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι με τα οποία συμφωνώ. Με μεγάλη επιφυλακτικότητα προσεγγίζω αυτό το σύμφωνο που υπέβαλαν οι Μέρκελ και Σαρκοζή. Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε πολύ καλά τα κίνητρά τους ε, είναι ε, ευφυείς στη στρατηγική τους. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι δεν έχουν κάποιο ε, λόγο που το υποβάλλουν και ότι δεν εννοούν αυτά που λέγουν. Άρα το θέμα σοβαρεύει. Εάν εννοούν την μέθοδο αυτή τη μαριθμοποίηση των τιμών είμαι πολύ επιφυλακτικός. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να θεωρηθεί και ως μείωση των συντάξεων ε, το φρένο στο δανεισμό ε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και έχουμε δει τα προβλήματα των χωρών Ελλάδα-Ιρλανδία. Είμαι επιφυλακτικός λοιπόν σε ό,τι αφορά την προτινόμενη αυτή επίλυση των προβλημάτων και περιμένω πάνω απ' όλα διαφάνεια. Ελπίζω, ε, ε, νομίζω ότι θα υποστηριχθείτε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν και εσεί ταχθείτε υπέρ τη μεγαλύτερη διαφάνεια. και αν τα φροντίστε τα παιχνίδια αυτά να μην γίνονται πίσω από την πλάτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν θέλουμε περικοπές πρέπει να το πούμε καθαρά. Όχι ε, μέσα από ε, να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα στόχο που δεν βρίσκει σύμφωνους όλους, ούτε εσάς κύριε Μπαρόζο. Συμφωνούμε για μια συντονισμένη οικονομική ε, πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση, μια ε, οικονομική διακυβέρνηση που θα αξίζει το όνομά της, που θα έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και που θα δημιουργήσει μια βιώσιμη ε, αηφόρο Ευρώπη. Επίσης είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε για τροποποίηση της συνθήκης. Ε, μέσα από μια κοινωνική ρήτρα πρόοδου. Περιμένουμε όμως ε, μια πιο έγκαιρη και ε, περιεκτική ενημέρωση και ένταξη του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες. Χωρίς ενημέρωση δεν μπορεί να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο τις διαδικασίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπίσκι. Και τώρα εξ ονόματος της Ευρώπης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για δύο λεπτά ο κύριος Φαράζ. Κύριε Παράσου, χάρηκα για τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τον κόσμο. Αλλά δεν ήταν αρκετά ηρωνικό. Μας είπατε για την ε, Αίγυπτο, για τις επαναστάσει, για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι όταν ψηφίζεις για κάποιον. Ξέρει τι κάνει και όταν δεν το θέλεις, τον πετάς. Και μετά φέρνει κάποιον άλλον που τον ψηφίζει και πάλι. Τι ηρωνία λοιπόν. Μα είπατε μετά, εν κρίση του ευρώ, πρέπει να ενισχύσουμε την κοινοτική μέθοδο, μα είπατε. Για εμάς που, για το κοινό που μας ε, βλέπει, η κοινοτική μέθοδος σημαίνει ότι προτείνονται κρυπτό και παραβεί στο νόμι από ανθρώπους σαν και εσάς. Ναι, ξέρω, ξέρω. Ναι, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας υπερψήφισε. Αυτά δεν είναι δημοκρατία, κύριε Μπαρόσο. Από τη μια μεριά μας λέτε ότι η δημοκρατία είναι καλό πράγμα και από την άλλη ε, ότι δεν είναι για την Ευρώπη. Και έχουμε και τον κύριο Φερχόφστατ το Βέλγιο, ο οποίο πιστεύει ότι όλα τα εθνικά κράτη πρέπει να καταργηθούν, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί και να συμβεί. Και μα μας λέτε, θέλουμε Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Κανεί δεν την υπερψήφισε, κανεί δεν μα ρώτησε αν τη θέλουμε. Εσεί, αν θέλετε, ψηφίστε τη. Αλλά οι λαοί τη Ευρώπη, κύριε Φερχόφστατ, δεν ψήφισαν για μια Οικονομική Ένωση. Τι θα συζητήσουμε λοιπόν την Παρασκευή, την Πορτογαλία, γιατί μετά από την διάσωση της Ελλάδας και της Ιρλανδίας είναι φανερό ότι οι αγορές στέλνουν το μήνυμα. Ελάτε, έρχεται το νούμερο 3, ήρθε το νούμερο 3. Η Πορτογαλία. Η... Τα επιτόκια των ε, πορτογαλικών ομολόγων είναι στο 7,6. Εκεί φτάσαμε. Και στο σημείο αυτό περίπου διασώθηκε και η Ιρλανδία. Και τον Απρίλιο, αν θυμάστε, είχαμε μια ε, εξαγορά πορτογαλικού χρέους που πρέπει τώρα να το ξαναδιασώσουμε. 80% του πορτογαλικού χρέου αγοράστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φτάνει πια, δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουμε να επαναγοράζουμε το δικό μας χρέος. Αν το κάνουμε αυτό, η επόμενη κρίση δεν θα αφορά κάποια χώρα, αλλά την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαράζ. Μια ερώτηση προς εσάς από τον Μάρτιν Σούλς. Τη δέχεστε? Παρακαλώ κύριε Σούλς. Κύριε Σούλς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υποθέτω ότι δεν το γνωρίζετε, αλλά θα σας ρωτήσω παρόλα αυτά. Πάντοτε αναφέρεστε στο Βέλγιο ως μη υπάρχον κράτος το είπατε και στον κύριο Φανρόπα και τώρα στον κύριο Φερχόφστετ. Γνωρίζετε πάνω σε ποια βάση έχει ιδρυθεί το βελγικό κράτος. Χαίρομαι που με ρωτήσετε. Το πρόβλημα είναι όταν δημιουργείς ένα τεχνητό κράτος που περιέχει πάνω από μία γλωσσική ομάδα, το Βέλγιο δηλαδή, και κατόπιν μπορείς για ένα χρονικό διάστημα να συγκρατήσει το κράτο αυτό, αλλά είτε μιλάμε για το Βέλγιο, τη Ιουγκοσλαβία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει τελείω διαφορετικέ γλώσσε και κουλτούρε, θα διαλυθεί. Και αυτό που σα ανησυχεί με το Βέλγιο και ενόχλησε πάρα πολύ τον κύριο Βανρόμπε και τον κύριο Φεχόστατ, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι το Βέλγιο είναι ένας μικροκόσμος ολόκληρου του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Εκτός μικροφώνου σχόλια και άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Διαπιστώνω ότι ο εκπρόσωπος ενός κόμματος ε, που είναι για την ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν γνωρίζει ότι το Βασίλειο του Βελγίου ιδρύθηκε μετά από πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ερώτηση αυτή. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση της γαλάζιας κάρτας, αν δέχεται ο κύριος Φαράζου και μετά θα ξαναγυρίσουμε στους ομιλητές. Ο κύριος Ντερόσα. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Ντερόσα. Μια ερώτηση από την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ελπίζω να μην προσβάλλει αυτό τον κύριο Φαράτζου. Είπατε και ξέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από του Άγγλου, του Σκοτσέζους, του Αλλού και του Βορειοϊρλανδού. Αυτό δεν είναι μια ένωση εθνών, παρακαλώ. Και μάλιστα υπερήφανων λαών. Καλή ερώτηση, λέει ο κ. Φάρατσου. Κύριε Σούλτ, έχετε δίκιο. Το Βέλγιο όντω ήταν ε, βρετανική εφευρεσία, αλλά και βρετανικό λάθο. Έχουμε κάνει πολλά λάθη ανά του αιώνε. Κάναμε καλά πράγματα, κάναμε και λάθο. Όπω, όπως ακριβώς και η χώρα σας, η Γερμανία. Η γερμανική ιστορία δεν ε, βρίσκει μόνο καλών πραγμάτων. Και το Ενωμένο Βασίλειο έχει κάνει πράγματα που προβλημάτισαν. Ιρλανδία, δείτε τι έγινε. Το 1921, δεν κάνω λάθος, απέκτησε η Ιρλανδία την ανεξαρτησία της. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσουμε μαζί διαφορετικά διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές κουλτούρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο τη Αγγλία, Ουαλία και τη Σκωτία δουλεύει προ το παρόν, ναι, γιατί υπάρχει συνένεση. Αν δεν υπήρχε συνένεση και είχαμε ζητήσει, είχαν ζητήσει δημοψηφίσματα, τότε αυτά τα έθνη ενδεχομένω θα διασπώνται και πάλι. Διακόπτη πρόεδρο. Κανεί όμω στην Ευρώπη δεν είχε αυτήν την ευκαιρία ακριβώ να ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ προτείνω να συνεχίσουμε με τους ομιλητές. Η κυρία Λεπέν δεν είναι παρούσα. Προχωρούμε στην κυρία Βόρτμαν Κόλ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Πρόεδρε, το Συμβούλιο πρέπει να, να αποκτήσει μεγαλύτερη φιλοδοξία για να, για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό. Καλό αυτό. Θα ήθελα ωστόσο να επανέλθω σε αυτό που αναφέρθηκε προς τον κύριο Μπαρόζη για τον τρόπο με τον οποίο ανέλαβε η Επιτροπή τα πράγματα σε ό,τι αφορά το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Και ο Μάρτιν Σούλτ σήμερα συμφώνησε επί του θέματος αυτού και πρέπει να το υπογραμμίσω. Συνεργαστήκατε με τον κύριο Βαν όμως υπάρχει ένα ολόκληρο νομοθετικό πακέτο που βρίσκεται επιτάπητο στο Κοινοβούλιο και εμείς είμαστε συνομοθέτες στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να θέσουμε τα πράγματα ε, με σαφή τρόπο. Το Κοινοβούλιο υπέβαλε 2.000 τροπολογίες. Εάν διαβάσουμε τις τροπολογίες αυτές θα δούμε μια σειρά θεμάτων συμφώνου σταθερότητα. Όλα αυτά, ε, τα γνωστικότητα, συγγνώμη, όλα αυτά απαιτούν μεγαλύτερη φιλοδοξία και αυτό που με ανησυχεί είναι πώς θα συνδέσουμε το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την στρατηγική 2020. Κύριε Μπαρόζο, θα χρησιμοποιήσετε πραγματικά το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής ούτως ώστε να υπάρξει σύνδεση μεταξύ του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας και του νομοθετικού πακέτου. Αν όχι, τι θα κάνει το κοινό. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να λάβει τον ρόλο του ως συνομοθέτη. Κυρία Φεραίρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έρχομαι από μια χώρα που υπάρχει ως ανεξάρτητη εδώ και οκτώ αιώνες. Παρά τα αυτά, σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα μπορέσει να συνομιλεί σε ισότιμη βάση με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Η κρίση που διανύουμε είναι μια κρίση της ζώνης ευρώ, της ευρωζώνης, διότι το ενίο νόμισμα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχει σοβαρή, μόνιμη ε, δουλειά σύγκλησης όλων των πλευρών που μετέχουν στο ενιονόμισμα νόμισμα. Όταν υπάρχει ωστόσο πραγματική ουσιαστική σύγκληση. Μέχρι τώρα εμείς ετοιμάσαμε δείκτες ονομαστικής σύγκληση μόνο, κάτι τελείως διαφορετικό. Επήγε λοιπόν η Ευρώπη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε και στον τομέα αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα στέρεο ταμείο ε, σταθερότητας που θα βοηθά και θα επιτρέπει τις χώρες σε δυσκολία να προχωρήσουν στη σύγκληση με αποδεκτά, όχι απαγορευτικά επιτόκια και χωρίς να χρειάζεται να περικόπτει στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις για να πετύχει μια τέτοια σύγκληση καθώς και για να μπορέσει να επιστρέψει αυτό που δανείστηκε σε κάποια στιγμή κρίσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν για να πετύχουμε αυτά μια δραστήρια Επιτροπή που θα μετέχει στην ε, διαχείριση αυτού του Ταμείου Σταθερότητας αλλά χρειαζόμαστε και ευρωομόλογα που θα ακού, ακούει τα μηνύματα που της δίνει σήμερα το Κοινοβούλιο μέσω νέων, νέων πηγών ιδίων πόρων για να φτάσει σε έναν προϋπολογισμό αποτελεσματικό και ουσιαστικό. Εμείς εγκρίναμε προηγουμένως την έκθεση υποδηματά που υποστηρίζει την ανάγκη να υπάρξει μια φορολογήση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία. Χρειαζόμαστε γι' αυτό ένα ισχυρό κοινοβούλιο, αλλά και μια επιτροπή ικανή όχι μόνο να αντιδρά, αλλά και να δρά, υιοθετώντα πρωτοβουλίε που είναι τόσο αναγκαίε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ακούστηκαν πολλά τα οποία συμμερίζομαι. Τρεις λέξεις όμως, επιτρέψτε μου. Η πρώτη είναι σεβασμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όντως συναποφασίζον όργανο, όχι που το θέλησε. Το θέλησαν οι κυβερνήσεις που συνυπέγραψαν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και γι' αυτό δεν δεχόμαστε να ενημερωνόμαστε για σημαντικές συζητήσεις οι οποίες αφορούν την διακυβέρνηση μέσω Google ή μέσω των αγγλόφωνων εφημερίδων. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο θα συζητήσω κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόσο και από τους εργάτες του κύριου Ρομπά είναι να μας σεβαστείτε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερη λέξη, δημοκρατία. Ποτέ δεν είδαμε από τον 18ο τουλάχιστον αιώνα ένα σύστημα με διαχωρισμό εξουσιών να προσπαθεί να αυτοκυρωθεί. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών. Υπάρχουν αυτοί που αποφασίζουν και αυτοί που ελέγχουν. Το Συμβούλιο είναι συνένοχος κύριε Παρόζο που προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα απόφασης. Και τρίτη λέξη, αποτελεσματικότητα και απόδοση. Εάν οι αποφάσεις χάνουν το περιεχόμενό τους, θα μείνουμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Και δέκα χρόνια μετά θα είμαστε εκεί πάλι στο μηδέν. Α κάνουμε λοιπόν τη δουλειά μα. Ζητούμε σεβασμό, θα περιμένουμε τη δημοκρατία αλλά και τη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Πόρτα. Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδε ο διεθνή τύπο σχολίαζε δηλώσει, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την πιθανότητα η Πορτογαλία να χρειαστεί να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το ερμηνεύεται αυτό ως παρακίνηση. Σας ερωτώ λοιπόν. Τρεις ερωτήσεις, ζητώ τρεις ειλικρινές απαντήσεις. Τι κερδίζει από το δούνο του η Πορτογαλία και από τον μηχανισμό σταθερότητας όπως είναι σήμερα. Δεύτερον, Ποιε είναι οι αλλαγέ που θεωρείτε εσεί απαραίτητε στον παρόντο μηχανισμό για να αποφύγουμε να ξανασυμβούν αυτά τα οποία έγιναν στην Ιρλανδία. Μείωση των μισθών, ε, απίστευτα ψηλά επιτόκια κλπ. Και τρίτη ερώτηση. Πώς περιμένετε ότι θα σας ξαναμπιστευτούμε όταν όλε οι υποφάσει συμπεριλαμβανομένων και αυτών τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τελικώς όλο και χειρότερε για τι φτωχέ χώρες και υπονομεύουν την ανάπτυξη. Ο κύριος Γκοζές, 1,5 λεπτό. Συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Γκουλάρ προηγουμένω για τα, τις αναγκαίες προϋποθέσεις που οδηγούν στο εξή. Ακόμα και αν καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρξει ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων, παρά τα αυτά είναι αναγκαία η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ω μόνη προπόθεση που θα επιτρέψει στου πολίτε, του οποίου εκπροσωπούμε, να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ένα συγκεκριμένο θέμα θα αναφέρω. Κάθε μέρα μα σπρώχνουν οι χρηματοοικονομικέ αγορέ, οι οποίε ε, συχνά περιλαμβάνουν ε, ε, εκπροσωπούνται νέους οι οποίοι πέρασαν από τα Game Boy στους κομπιούτερς χωρίς να το σκεφτούν και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τις χώρες να τρέμουν. Αν θέλουμε να ελέγξουμε τις αγοράς δεν θα το κάνουμε καταργώντας τις αγορές. Δεν θέλω, δεν είναι ανήκω στην ομάδα που θέλει την κατάργηση της αγοράς. Αλλά τι θέλουν οι αγορές. Θέλουν την αποφυγή του κινδύνου. Το παιχνίδι στην αγορά είναι να περάσει τον κίνδυνο σε κάποιον άλλον Ούτω ώστε κανείς συναλλασσόμενο δεν είναι ικανοποιημένο όσο υπάρχει κίνδυνο. Εμεί λοιπόν θέλουμε να επαναφέρουμε την ισορροπία στην χρήση μεταγορέ, να δώσουμε σαφεί γραμμέ, να μην περνάμε του χιλιάδες ιδέες που δεν υλοποιούνται. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να ελέγξει αυτή τη χρηματοοικονομική διάσταση, κάτι αναγκαίο για τις χώρες μας. Πρέπει για να το πετύχουμε αυτό, και εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δώσουμε σαφή ορίζοντα, σαφή μέτρα και ξεκάθαρη αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά τον καλό οικονομικό συντονισμό. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Ντερόσας για 1,5, Ντερόσα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η θελημένη αποφυγή της οικονομικής διακυβέρνησης και ένας κανονισμός ε, για τις, και ενός κανονισμού για τις τράπεζες μας έφερε σε αυτή την ε, ε, κρίση. απώλεια συντάξεων, θέσεων εργασίας είναι γνωστά. Πρόεδρε Μπαρόσο, Επίτροπε Όλη Ρεν, θα πρέπει να με πείσετε ότι η οικονομική διακυβέρνηση είναι στα σχέδιά σας και ότι θα έχει στέρεες βάσεις. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να πείσετε για την αναγκαιότητά της τους λαούς της Ευρώπης αποδεικνύοντας την ομιμοποίησή της, ε, απορρίπτοντας ε, προτάσεις που δεν ε, βασίζονται στη συνθήκη και στην κοινοτική μέθοδο. Θα πρέπει να μην είναι προς το συμφέρον δύο, τριών, τεσσάρων οικονομικά ισχυρών κρατών. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ένωσης αυτό που θα συμφωνηθεί στην άτυπη σύνοδο της 11 αυτό που θα συμφωνηθεί εκεί λοιπόν, θα μπορεί να βρει σύμφωνη την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Η Ιρλανδική κυβέρνηση που εξελέγει πρόσφατα έχει ισχυρή εντολή στην Ιρλανδία και παραθέτω από το πρόγραμμα που συμφώνησαν ε, πριν από λίγο. Θα πρέπει να ε, αποφύγουμε την ε, αφαιρεγγιότητα ως κράτος θα πρέπει να αντιστρέψουμε την αποτυχία ε, ε, αντιμετώπισης της ε, οικονομίας στην Ιρλανδία. Και, αν μου επιτρέπετε, διακόπτη πρόεδρος. Τελειώνω. Μία φράση μόνο. Συμβάλλει στην ε, ευρύτερη δημοσιονομική αστάθεια στην ε, ζώνη του ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ διακόπτη τον κύριο Ντερόσα, η πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Σαρόν Μπόλς για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, κάθε εβδομάδα ο τύπος είναι γεμάτος πληροφορίες για άλλες καινούργιε ή αλλαγμένε προτάσεις από μια χώρα, από το Συμβούλιο, από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Συγχαίρω τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας διότι πραγματικά ε, πρόσεξε τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου και αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα και την πορεία που θέλουμε να δώσουμε. Το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας είναι ένα βασικό παράδειγμα. Ήδη υπάρχει μια σειρά ενδιαφερουσών ινδεών στην τροποποίηση μας για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά δεν θα έχουμε δυσκολία να προχωρήσουμε σε συναπόφαση για να συγχωνεύσουμε την έκβαση των αποφάσεων μεταξύ Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επιλέγουμε πράγματα από την ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά δεν είναι απ' έξω ένα φρούριο και ένα ισότιμος χώρος ε, συνεργασίας εσωτερικό. Είναι μια προσφορά ανταγωνιστικότητας και ένα μείγμα για την επίτευξη της ανάκαμψης και για την οικονομική διακυβέρνηση. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα μόνιμο μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθερότητας που θα στηρίζεται σε χρονια, που θα έχει χρονική, ευρύ χρονικό ορίζοντα και θα στηρίζεται σε συγκεκριμένε προτεραιότητε. Προ του Γερμανού που ανησυχούν για την ε, χρηματοδότηση τη διαδικασία αυτή, θα σα πω, δείτε τι ζητά η τράπεζά σα. Ανακεφαλαίωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών. Οι γερμανικέ τράπεζε θα, θα, πάρω, θα κάνουν 10 χρόνια για να αναγνωρίσουν τι σημείε ε, ε, το, τις ζημίες τους ακόμα και σε κρατικά χρεόγραφα. Η μεταφορά λοιπόν, στη, η μεταφορά κονδυλίων στις γερμανικές τράπεζες θα πρέπει και αυτό να σας ανησυχεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μηχανισμούς όπως αυτούς του μόνιμου μηχανισμού. Για τα επιτόκια πρέπει να υπάρξει εξισορροπία ισορροπία μεταξύ ε, αντοχής και κινδύνου. Διακόπτεται εν τέλει η διακόπτη η πρόεδρος. Δεν... Έχετε κατά πολύ υπερβεί το χρόνο σας. Και τώρα ο κύριο Φέιο, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, οι δύσκολοι καιροί απαιτούν θραλές αποφάσεις. Γι' αυτό είμαστε και εδώ. Γι' αυτό συγχαίρω τον πρόεδρο Μπαρόσο για τις ιδέες που κατέθεσε εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει και αυτό σαφή θέση με τη μορφή εκθέσεων για το ευρώ, για την ανάγκη σταθερότητας, την ανάγκη διαχείρισης του ευρώ, την ανάγκη ανάπτυξης. Η κατάσταση έχει πολλές πτυχές. Το ταμείο και οι μηχανισμοί αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των χωρών που πληρώνουν υπερβολικά υψηλά επιτόκια για το χρέο του. Μια άλλη πτυχή είναι η ανταγωνιστικότητα για την οποία πρέπει να κάνουμε κάτι. Χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική πολιτική η οποία θα συμβάλλει στην εξασφάλιση επενδύσεων. Το θέμα είναι λοιπόν η δημιουργία πλούτου στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε πιο ευρωπαϊκού θεσμού, πιο ευρωπαϊκέ προσεγγίσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε σαφεί αποφάσει και τι ανακοίνωσε. Ω όφιλε, όχι μόνο για τα μέσα, δεν είναι καιρό για ιδεολογήματα. Α μην ξεχνούμε του πολίτε μα. Χρειάζονται αποφάσει σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στη διαδικασία κάτω στη ΆΗ τώρα. Δεν εκπλήσει ότι το ενδιαφέρον είναι ζωηρότατο. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Θα δώσω το λόγο σε έξι συναδέλφους μόνο και από την αρχή το λέω για να είστε προετοιμασμένοι. Είναι ο κύριος Τάουτς Βόλς, η Γουαλτιέρη, Γκάλαχερ, η κυρία Φιγκερέιδο, Πάσκα και ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ο κύριος Σάρους Φόλσκι, παρακαλώ, έχετε πρώτο το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η κρίση της Ευρωζώνης, αλλά των δημοσίων οικονομικών κρατών μελών που ήταν ε, στην Ευρωζώνη. Ε, θα μπορούσε να είναι η ε, Ουγγαρία. Γιατί θα πρέπει να δημιουργούμε ε, αδικαιολόγητες διαχωριστικές γραμμές. Γιατί να δημιουργούμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Εσείς κύριε Μπαρόζο είστε θεματοφύλακες της συνθήκης. Γιατί αποκλείονται οι πρόθυμοι και οι ικανοί. Ε, γιατί θα πρέπει να βαθαίνει ε, η διαφορετική να βαθαίνουν οι διαφορές στις δημοσιονομικές μας πολιτικές τα 27 κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ηγέτες των 27 και όχι ε, οι εκπρόσωποι μόνο μιας περιορισμένης ομάδας χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Μπαχέρη. Ευχαριστώ. Χθε στην Συνταγματική Επιτροπή ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ε, μεταρρύθμιση της συνθήκης για τη θέσπιση του μηχανισμού σταθερότητας το κείμενο προτείνει μια αλλαγή στην ε, πρόταση τροποποίηση συνθήκη τη Λισαβόνα ε, που καθορίζει μια διαδικασία που διαφυλάσσοντα τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του Ταμείου δικαιολογεί την συμπερίληψη του κανόνα αυτή στη συνθήκη, του αυτού στη συνθήκη και περιλαμβάνει σαφεί προτάσει για τη λειτουργία του μηχανισμού, τόσο ώστε να είναι συμβατό με τι ευθύνε που αναφέρει η συνθήκη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την απέτηση πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης που αν ήταν, αν ήταν διακυβερνητική δεν θα λειτουργούσε απλά και μόνο. Για να επαναφέρω μια μεταφορά που χρησιμοποίησατε εσεί ε, κύριε Πρόεδρε στην προηγούμενη συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να τοποθετηθεί αυτό το διακυβερνητικό βαγόνι σε σιδηροτροχέ και σε τρένο τη Ένωση, αναφέροντα στην Επιτροπή το ρόλο που τη αρμόζει στη διαχείριση αυτού του ε, τρένου. Πώ βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτάσει του Κοινοβουλίου και είναι έτοιμη να συμβάλλει στι διαπραγματεύσει, Διακόπτεται ο μιλητής. Ευχαριστώ. Κύριος Γκάλαχερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η λαδιά είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία με ισχυρή συγκέντρωση αμέσων ξένων επενδύσεων. Το ποστό του φόρου, δελεστής του φόρου, είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Αντί λοιπόν να αυξήσουμε τους ε, φόρους, ας κοιτάξουμε να κρατήσουμε αυτές τις ψηλού επίπεδου εταιρείε στην Ιρλανδία. Κάθε ισοπαίδωση, κάθε εναρμόνιση των, των φορολογικών συντελεστών στην Ευρώπη θα βλάψει την Ιρλανδία και τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να πετυχαίνουμε ανάκαμψη. Ας μην ξεχνούμε ότι η Ιρλανδία, όπως και άλλες μικρές χώρες, γεωγραφικά και ιστορικά είναι χώρα περιφερειακή ως προς την Ευρώπη. Οι χαμηλοί φόροι λοιπόν είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση των οικονομικών περιορισμών που προκύπτουν λόγω της θέση μας. Και ρωτώ τον Πρόεδρο, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βάσει της συνθήκης η φορολογική πολιτική παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέιδο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα, σήμερα γιορτάζουμε την ε, ημέρα της γυναίκας και ακούσαμε ωραία πράγματα για τα δικαιώματα των γυναικών. Τα οικονομικά ε, συμφέροντα βλέπουμε όμως σήμερα να ε, κυριαρχούν στην οικονομική διακυβέρνηση και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των χωρών και τις μεγάλες οικονομικές ε, διαφορές και δυσκολίες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό που θα αναμένουμε λοιπόν από το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας είναι επιδείνωση όλων των υφισταμένων προβλημάτων. Σημαίνει επίσης όμως ότι οι λαϊκοί αγώνες θα πρέπει να συνεχιστούν. Όπως είδαμε και στην Πορτογαλία και ε, στο παρελθόν και στο άμεσο μέλλον και το επόμενο ε, Σαββατοκυριακό. Αυτό ε, θα πρέπει να αναμένουμε από τις προτινόμενες αλλαγές. Σε τέτοιες εξελίξεις ελπίζει η Κομισιόν. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπη. Καταρχήν θα ήθελα να Ε, πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με βάση συγκεκριμένες και ηθελημένες αποφάσεις ε, των κρατών μελών ε, ούτως ώστε να συντονίζονται επελεγμένες αρμοδιότητες. Ελήφθη απόφαση για παραχώρηση μέρους της κυριαρχίας. Αν αποφασιστεί η οικονομική διακυβέρνηση σε επίπεδο ένωσης αυτό θα πρέπει να είναι μία απόφαση ε, γενικότερη με όλους τους εμπλεκομένους, όχι απόφαση των Βρυξελών. Όταν μιλάμε για συμφωνία κυρίαρχων κρατών, ε, τότε θα είναι μία ελεύθερη ε, απόφαση. Επίσης είναι σημαντικό να ενισχυθεί η στενότερη συνεργασία με πρωτοβουλίες από την Ευρωζώνη που βέβαια επέλεξε το κοινό νόμισμα. Μην αυτά πατώμεθα όμως κυρίες και κύριοι. Εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικούς κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Danke, Vorsitzende, insbesondere Ευχαριστώ πολύ και για την ε, δικαιοσύνη στη διαδικασία. Η ρύθμιση για την δημοσιονομική ε, πολιτική της Ένωσης ε, προβλέπει περαιτέρω βήματα προς την οικονομική διακυβέρνηση και βέβαια παρέμβαση και στην φορολογική στην κυριαρχία των κρατών μελών. το η τροποποίηση του άρθρου 136 ε, θα μπορούσε να οδηγήσει στην έγκριση των προτάσεων ε, Μέρκελ-Σαρκοζή. Τα, ε, οι χώρες της Ευρωζώνης μπορεί να συνεχίσουν να υφίστανται πιέσεις. αυτό θα οδηγήσει σε ε, ανατροπές σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαρόζο τι γίνεται με τις δεσμεύσεις ε, σχετικά με την ίση κατανομή των βαρών. Ε, με τις ε, πρόσφατες προτάσεις θεωρώ ότι όλα αυτά διακυβεύονται. Ευχαριστώ. Και για να κλείσουμε τη συζήτηση, ο κύριος Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καταρχάς, επειδή υπήρξαν συγκεκριμένα ερωτήματα για την Πορτογαλία, θα απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα η, εάν χρειαστεί να προσφύγει η Πορτογαλία στο μηχανισμό σταθερότητας ή όχι. Η απάντησή μου είναι ότι αυτό θα, απο, εξαρτηθεί από τι αποφασει των πορτογαλικών αρχών. Είναι ένα πρόβλημα κρατικού χρέους ε, της ε, Πορτογαλίας. Η προσφυγή στη βοήθεια ε, επινοήθηκε ω έσχατη λύση. Αν μια χώρα μπορεί, θέλει να αποφασίσει να προσφύγει, μπορεί να το κάνει αλλά υπάρχει και κόστος ε, αν ε, προσφύγει κανείς σε αυτό το ταμείο. Αν μια χώρα λοιπόν μπορεί να το αποφύγει, τόσο το καλύτερο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τούτο είναι μια απόφαση των εθνικών αρχών. Αν θέλουν ή όχι να προσφύγουν ε, στο ταμείο αυτό ή να υποβάλουν έτοιμα να προσφύγουν στο ταμείο αυτό. Κατόπιν, αυτό που θα ήθελα να δω στο τι θα ήθελα να έχει αυτό το ταμείο. Το δεν είναι θέμα τι μ' αρέσει εμένα και τι δεν μ' αρέσει. Είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις χώρες της Ευρωζώνης, ούτως ώστε το, ο μηχανισμός αυτός να έχει ενισχυμένη ικανότητα ε, χρηματοδότησης για να είναι και να, και να έχει μεγαλύτερη ευελιξία. Υπάρχουν κάποιες ευαίσθητες διαστάσεις σε επίπεδο αγορών, γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι φρόνιμο να σας προαναγγείλω τις προθέσεις μας που δεν είναι συγκεκριμένες και δεν έχουν καθοριστεί. Πάντως δουλεύουμε σε επίπεδο χωρών Ευρωζώνης και η Επιτροπή στην αξιολόγηση, την ετήσια αξιολόγησή τη για την ανάπτυξη παρουσίασε σαφεί προτάσει για να ενισχύσει το ταμείο αυτό και να διευρύνει τι δραστηριότητε του. Τώρα, το κατά πόσον η πολιτική αυτή θα έπρεπε ή θα μπορούσε να αλλάξει. Εγώ πιστεύω πως όχι. Θα ήταν, ε, δεν θα ήταν υπεύθυνο χώρες με ε, οι χώρε με ιδιωτικό και δημόσιο χρέο δεν πρέπει να μειώσουν τι προσπάθειε εξυγίανση του προπολογισμού και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όταν μια χώρα έχει τόσο υψηλό χρέο, θα πρέπει να, ανακτήσει την εμπιστοσύνη τη αγορά η οικονομική τη κατάσταση δεν μπορεί να να, είναι σταθερή. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις πλέον ευάλωτε χώρες δεν θα πρέπει να έχουμε μια ουτοπιστική προσέγγιση αλλά να, να υποστηρίξουμε τις προσπαθίες τους για να εξηγιάνουν τον προπολογισμό τους και να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των αγορών. Βεβαίω, δεν ε, μπορεί να κάνει κάθε χώρα πολλά πράγματα μόνη τη. Χρειάζεται μια συλλογική κοινή προσπάθεια των χωρών τη Ευρωζώνη και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Προφανώ η Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε για να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Η Επιτροπή ωστόσο προτείνει αλλά για τα ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας, την προσφυγή ή για θέματα εκτός συνθήκης όπως το Ταμείο, η απόφαση είναι απόφαση των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Να σας πω το εξής. Προφανώς οι πολλοί, πολλές επικρίσεις από τους ομιλητές ήταν επικρίσεις προς κυβερνήσεις. Δεν μιλάω εγώ εξ ονόματός τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο προτάσεων οικονομικής διακυβέρνησης. Δοκιμάσαμε τα όρια της φιλοδοξίας των κυβερνήσεων και το πακέτο διακυβέρνησης που παρουσίασε ο κύριος Ρεν και εγώ και το πακέτο αυτό δεν θέλησαν να το δεχθούν τα κράτη-μέλη, να δεχθούν το επίπεδο αρχικών ε, φιλοδοξιών. Εμείς υποβάλαμε και νομοθετικές προτάσεις. Τώρα, μια νέα ιδέα που προτάθηκε, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό. Προσπαθούμε να περάσουμε όσο περισσότερο γίνεται το πακέτο αυτό, να του βάλουμε όσο περισσότερο γίνεται ε, κοινοτική διάσταση. Σας το λέω ειλικρινά. Εμείς προσπαθούμε να είναι χρήσιμη η ιδέα αυτή, να έχει ε, ε, προστιθέμενη αξία και για την απασχόληση και ανάπτυξη που παραμένει όπως είπα προτεραιότητα της Επιτροπής και για την ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης. Δεν χρειάζεται να μας θυμίζετε ότι είμαστε θεματοφύλακες της συνθήκης. Το δείξαμε και το δείχνουμε συνεχώς για θέματα εσωτερικής αγοράς, ανταγωνισμού, μη διάκρισης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω εκ νέου ότι η Επιτροπή δεν θα διστάσει να προσφύγει σε κάθε μέσο αν θεωρεί ότι υπάρχουν αρχές ή κανόνες της συνθήκης που αμφιτέθεται επαμφιβόλο από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλου οργάνου. Γι' αυτό η κανονες στις συνθηκες που αμφιτεθεται επαμφιβολο απο αποφασεις του ευρωπαικου συμβουλιου η οποιοδηποτε αλλου οργανου γι αυτο η δουλεια μας είναι μακρόπνοη, σοβαρή με και γίνεται με αίσθημα ευθύνης. Διότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά λεπτή στιγμή. Σε μια στιγμή όπου πολλές κυβερνήσει το πρώτο πράγμα που κοιτούν το πρωί, που ξυπνάνε είναι τι γίνεται με την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους. Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν είναι αδιάφορο. Η, αυτό που δημιουργούμε δεν είναι αδιάφορο. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σαν Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όταν κάνουμε προτάσεις γνωρίζοντας ότι πρέπει να έχουν ε, στόχο να υλοποιηθούν και να μην είναι μόνο ωραίες αναγγελίες και μετά να δημιουργούν απογοήσεις. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, να αυξηθούν οι ε, να διαιρεθεί η Ευρωζώνη ή να διαιρεθεί η Ένωση. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα τηρεί πάντα τους στόχους της μέγιστης φιλοδοξίας και να επιθυμεί τη συμμετοχή του του Κοινοβουλίου στο Σύμφωνο Λογονιστικότητας. Η Επιτροπή θα πει στις κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να διατηρούμε ένα ρόλο. Όχι επειδή είμαστε εγωιστές θεσμικά. Ε, αλλά διότι πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτροπή και η κοινοτική μέθοδος είναι εγγύηση αποφυγής των διαιρέσεων μεταξύ Ευρωζώνης και Λυπής Ένωσης για να αποφεύγονται επιθέσεις στην ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς και εξασφαλίζει την αποφυγή χρησιμοποίησης άλλων μηχανισμών όπως του Συμφώνου Σταθερότητα και της Ανάπτυξης. εγγύηση ότι μένουμε Ευρωπαίοι με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ήμουν ειλικρινέστετος, ανοιχτός, με διαφάνεια. Και σας το ξαναλέω, κάνει η Επιτροπή τη δουλειά της με επικοδομητικό τρόπο, προσπαθώντας να διασώσει μια ιδέα που αν παρουσιάζεται με σωστό τρόπο θα μπορέσει να συμβάλλει στις προσπάθειες διακυβέρνησης. Το υπογράμμισαν αυτό κάποιοι από εσά. Οι προσπάθειες για έναν συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ήταν πάντα στόχος της Επιτροπής και της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Αν θέλουν τώρα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε αυτό το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και σε κάποιου τομεί που μέχρι τώρα θεωρούνται εθνική αποκλειστικά αρμοδιότητα, αυτό πρέπει να το καλωσορίσουμε. Εφόσον βέβαια τούτο προσφέρει στην ανάπτυξη και την απασχόληση και εφόσον τηρείται το σύστημα κοινοτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το ζήτημα. Πιστεύω ότι η συζήτηση ήταν χρήσιμη και νομίζω ότι το μήνυμα του Κοινοβουλίου πέρασε στο Συμβούλιο. Ο πρόεδρος Μπούζεκ στην τελευταία παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρασε το, τη θέση του Κοινοβουλίου και Κοινοβούλιο και Επιτροπή πιστεύω θα είναι αποφασιστική στην υποστήριξη της κοινοτικής προσέγγισης ως μόνο τρόπο να πετύχει η Ευρώπη τους στόχους τους στόχους και της Ευρωζώνης και της σταθερότητας και της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλη την Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. ολοκληρώνει Και το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έκθεση προόδου 2010 σχετικά με την Τουρκία.